Madame la Présidente. La séance est reprise. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σύνοδο. Οι αρμόδιες αρχές της Λετωνίας είπαν ότι εξελέγει η κυρία Λιεπίνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικαθιστώντας τον κύριο Ντομπρόφσκι και αυτό από τις 19 Μαρτίου 2009 ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού